επόμενο θέμα Γκάμπια ε, θα δώσω το λόγο για 1,5 λεπτό τώρα στο λόγο, ε, τον λόγο στον κύριο Σεμπαστιά Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ψήφισμα με τόσο ευρία υποστήριξη στο Κοινοβουλίο μας. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Γκάμπια, η έλλειψη δημοκρατίας, ο κίνδυνος δίωξης και κράτησης και βασανιστήριων που υφίστανται πολλοί πολίτες της χώρας αυτής θα πρέπει και ειδικά ομάδων όπως η ΛΟΑΤ σημαίνουν το Κοινοβουλίο μας θα πρέπει να πάρει μια σαφή θέση καταγγελίας αυτών των φαινομένων. Μας φαίνεται ότι είναι ουσιώδες να περιλαμβάνεται σε αυτό το ψήφισμα και μια έκκληση για δράση της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Γκάμπια. Επίσης και μια έκκληση προς την ε, Ένωση, την Οικονομική Ένωση της Δυτικής Αφρικής και την Ένωση Αφρικανικής Ενότητας για να συνεχίσουν την καταγγελία των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ουσιώδες επίσης να παγώσει κάθε μορφή υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πρόεδρο Γιαμέ, ο οποίος έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανεκτό. Και φυσικά με την ε, εξαίρεση της ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί δεν μπορεί να πλήτεται ο λαός της Γκάμπια από τέτοια μέτρα. Έχουν έρθει 15.000 <clears throat> ετούντε άσυλο από την Κάμπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015. Καταλαβαίνετε τι αποστάσεις χρειάστηκαν να διατρέξουν και πόσα βάσανα έχουν περάσει για να μπορέσουν να φτάσουν εδώ. Δεν χρειάζονται περισσότερα στοιχεία. Θα πρέπει να δράσουμε τώρα για να σταματήσουμε αυτή την, αυτά τα βάσανα των ανθρώπων αυτών. Ο κύριος Κοράγια, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Διοικείται από έναν δικτάτορα η χώρα αυτή που έχει καταστρέψει τη δημοκρατία. Από το 1994 που ανέβηκε στην εξουσία μετά από ένα πραξικόπημα το μόνο που έχει δώσει στη χώρα είναι η διαφθορά και η ανελευθερία. Βασιλεύει ο φόβος, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων όπως και των ομοφιλοφίλων, και παρόλα αυτά φωτογραφίζεται ο πρόεδρος δίπλα από τον Ομπάμα και αγνοείται, αγνοούνται τα θύματα του στιγνού αυτού δικτάτορα. Πρέπει λοιπόν η Γκάμπια να επικυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών εναντίον των βασανιστήριων και να πάρει επιτέλους τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να σταματήσουν τα μέτρα τα οποία παίρνει βάρος των ομοφιλοφίλων στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Θα παρακαλώ να μιλάτε πιο αργά από εδώ και πέρα. Κύριος Δεμεσμάκερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει, ε, εκτός από αυτό που βλέπουν οι τουρίστες, ε, ένα άλλο πρόσωπο στην Κάμπια, ο οποίος γνωστός δικτάτορας ε, κυβερναϊκή, ο Τζαμέ πώς μπορεί κανείς να μιλήσει. Έχουμε τις μυστικές υπηρεσίες οι οποίες σπείρουν τον τρόμο στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, στα χωριά και ακόμη και τη, όχι απλά οι δημοσιογράφοι αλλά και οι ε, περί το Προέδρο είναι θύματα, τους κυνηγούν σαν θύραμα. παραβίασε πέρυσι το Σύνταγμα της χώρας κηρύσσοντας ε, τη χώρα Ισλαμική Δημοκρατία ο πρόεδρος, όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει ε, πολύ πιο προσεκτικά την κατάσταση στη μικρή αυτή αφρικανική χώρα ε, και ένα πρώτο βήμα θα ήταν οι ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές. Ευχαριστώ. Βασιλεύει ένα κλίμα φόβου στην Κάμπια και πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού προσπαθεί να μεταναστεύσει. Είναι μία από τις έξι πρώτες χώρες, ποσοστιαία βέβαια, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες που προσπαθούν να προστατευθούν στην Ευρώπη. Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων λοιπόν των, των μη κυβερνητικών οργανώσεων συνεχίζονται όπως επίσης και η απάνθρωπη συμπεριφορά από πλευρά των εκπροσώπων του καθεστώτος εις βάρος των πολιτών, όπως τα βασανιστήρια. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να συνδέσουμε την οικονομική βοήθεια με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας να παρακολουθήσουμε την κατάσταση στον τομέα ε, των σοφρονιστικών στη χώρα αυτή, όπως επίσης ε, και την συμπεριφορά της κυβέρνησης στις ομάδες των ομοφιλοφίλων. Η κυρία Σένρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Γκάμπια είναι μία από τις μικρότερες και φτωχότερες αφρικανικές χώρες. Η φτώχεια είναι γενικευμένη, κυριαρχεί στις αγροτικές περιοχές και οι γυναίκες βέβαια πλήττονται περισσότερο από αυτή την κατάσταση, όπως επίσης είναι και αυτές που παράγουν το 40% του συνόλου της γεωρικής παραγωγής, χωρίς όμως να ελέγχουν τις γιές, ούτε και να έχουν κάποιο ρόλο στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Ο ιός του έμπολα επίσης είχε 100 βεστημάτων, έπληξε και την τοπική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έδινε 14,2 εκατομμύρια, το 14 τα ανέστηλε αυτά τα χρήματα και φέτος το 31% των εσόδων της χώρας ε, θα ε, καταβληθούν για την αποπληρωμή του χρέους. Απαιτούμε η κυβέρνηση της Γκάμπια να θέσει ένα τέλος ε, στην καταστολή και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της θα πρέπει να συνεισφέρει ώστε ο λαός της Γκάμπη και ιδίω οι γυναίκες να βγουν από αυτή τη χρόνια αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ένα λεπτό τώρα ο κύριος Τζεχόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κάμπια δεν είναι η μόνη χώρα της Δυτικής Αφρικής όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι σε κίνδυνο. Η κατάσταση στη χώρα αυτή επιδεινώνεται εδώ και πολύ καιρό. Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταπατηθεί. Η ελευθερία της έκφρασης έχει καταπατηθεί. Έχουμε αυθαίρετη κράτηση σε φυλακές και απάνθρωπη μεταχείριση και βασανιστήρια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε πια καθόλου για αστικές ελευθερίες. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω απόλυτα την ανάγκη να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μειωθεί η οικονομική υποστήριξη προς την Γάμπια και επίσης θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση της Γάμπια να αντιμετωπίσει αυτή την πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γάμπια θα πρέπει να παρακολουθεί από κοντά τα, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων <clears throat> δικαιωμάτων και θα πρέπει να έρθει σε διάλογο με την αντιπολίτευση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται συνέχεια. Επόμενος ομιλητής. Κύριε Βάιτμαν, σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό περιλαμβάνει πολλές αντιφάσεις, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι. Η Γκάμπια θέλει να προσελκύσει τουρίστες, αλλά αναγκάζει το λαό της να αποχωρήσει από εκεί. Και ιδίως οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας μακρός κατάλογος παραβιάσεων που έχει λάβει η χώρα στην Κάμπια. Δεν υπάρχει το δικαίωμα του συναθρίζεστε ειρηνικά. Πολλές φορές οι διαδηλώσεις αντιμετωπίζονται με ακραία βία. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι καθώς και οι εκπρόσωποι της κοινότητας στο ΛΟΑΔ μπορούν να συλληφθούν αυθαίρετα και να βασανιστούν. Διατηρεί ένα κλίμα φόβου και καταπίεση η κυβέρνηση στην Γάμπια. Γι' αυτό χρειάζεται πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παραμείνει στην επικαιρότητα το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση θα πρέπει να κάνουν όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να υπάρξει η δημοκρατική διαδικασία στη χώρα αυτή. Μπορεί να φαίνεται μια χώρα ιδανική για τουρίστε, αλλά δεν είναι για του πολίτε τη. Ο κ. Βέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Γκάμπια είναι μία από τις 15 φτωχότερες χώρες του κόσμου εξαρτάται από τη διεθνή βοήθεια αλλά και την ενωσιακή βέβαια. Δεν υπάρχει όμως σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό και περιέκοψε δραστικά αυτή τη βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι το 1 τέταρτο του πληθυσμού της χώρας θα πεινάσει. Είχαμε εκλογές το Δεκέμβριο. Ο πρόεδρος ε, Τζαμέ ε, μάλλον θα υπάρχουν εκλογές και θα προσπαθήσει για πέμπτη φορά να επανεκλεγεί ο πρόεδρο. Οι αρχέ ε, ήδη απειλούν την αντιπολίτευση και του ε, πιθανούς υποψηφίους ε, και συλλαμβάνουν δημοσιογράφους και υπερμάχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. διώκουν στους πολιτικούς του αντιπάλου. Είχαμε τραγικά γεγονότα στις ειρηνικές ε, πρόσφατες διαδηλώσει σε Ρεκούντα. Πρέπει να συσταθεί μια ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή για να γίνουν δίκαιες εκλογές. Ευχαριστώ, David Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, υπάρχουν κάποιοι υπήκοοι τη Γκάμπια που ζουν στη δική μου εκλογική περιφέρεια, έχουν φύγει ε, για να γλιτώσουν από το στιγνό καθεστώς της χώρας ε, στο κατακεφαλήν, αν θέλουμε να υπολογίσουμε το κατακεφαλήν ποσοστό, υπάρχουν περισσότεροι μετανάστες από την Κάμπια, ακόμη και από τη Συρία. Αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, ιδίω αν λάβουμε υπόψη το ότι επειδή είναι πολύ μικρή η χώρα, μπορεί να είναι σε απόλυτα νούμερα μικρή αριθμή, αλλά σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τη χώρα είναι τεράστια. Υπήρχαν ε, κάποια εκατομμύρια ε, βοήθειας του 14 τα οποία ε, δεν δόθηκαν αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει διαβούλευση στο άρθρο 6 και αν δεν απελευθερωθούν εκτεβιστές οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από ειρηνικές διαδηλώσεις τους αν δεν σταματήσουν οι βεότητες ε, και τα βασανιστήρια, ε, θα πρέπει ε, να στείλουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να παρέχουμε βοήθεια, γιατί αφού είναι βίαιο και ομό το καθεστώς, σε τέτοια πρέπει να είναι και απάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπεθέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Γιούροβα, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για το κατεπήγον αυτό ψήφισμα. Είναι πληρέστατο ε, για την Κάμπια, να το ψηφίσουμε σε λίγο. Δυσκολεύομαι όμως να πιστέψω ότι ένας δικτάτορας που πάνω από 20 χρόνια είναι στην εξουσία και απειλεί ότι θα αποκεφαλίζει τους ε, ομοφιλόφιλους και που ε, προσπαθεί με κάποια φυτά ε, να θεραπεύσει έτσι και τα λοιπά πρέπει να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό που πλήττεται. Ε, όπως είπα με και προηγουμένως άλλοι συνάδελφοι, από τις 15 φτωχότερες χώρες είναι η Γκάμπια. Έχουμε επίσης ε, αυθαίρετες προσοχές συλλήψεις, δολοφονίες, βασανιστήρια. Όλα αυτά κάνουν ε, την χώρα ένα πρόβλημα. Έχει γίνει και παράδοση σεξουαλικού τουρισμού μεταξύ άλλων. Πιστεύω ότι και με τις εκλογέ ε, φέτος ε, πολλές χιλιάδες ε, κάτοικοι θα βγουν στους δρόμους. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε είτε να στείλουμε μια αποστολή παρατήρησης είτε κάπως μέσω της ομάδας στήριξης της Δημοκρατίας και εκλογικού συντονισμού να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγγίλη για ένα λεπτό. Κι εγώ ενοχλούμε πάρα πολύ και ανησυχώ για την κατάσταση στην Κάμπια γιατί η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει με βία και έχει συλλάβει ειρηνικούς διαδηλωτές, έχουν ε, βασανιστεί και ένας ακτιβιστής πέθανε ενώ ήταν σε κράτηση. Όλα αυτά γίνονται ενώ συγχρόνως γίνεται απόλυτη παρενόχληση και καταπίεση αγοριστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και εκπροσώπων της κοινότητας των ΛΟΑΔ. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει 8 εκατομμύρια σε βοήθεια, να ασκήσει πίεση προς την Γκάμπια, ώστε να ε, αναστείλει την νομοθεσία που έχει κατά τον ΛΟΑΔ. Οι αρχές της ε, Γκάμπια όμως θα πρέπει να καταλάβουν δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις κάτω από τέτοιες συνθήκες. <clears throat> Θα πρέπει όμως να πάρουμε μια ηγετική στάση, να εργαστούμε μαζί με την Αφρικανική Ένωση και μαζί με την αντιπολίτευση. Εγώ ανησυχώ και για τις εκλογές που θα γίνουν τον Δεκέμβριο. Μπορούν να γίνουν πραγματικά ελεύθερες εκλογές τον Δεκέμβριο κάτω από τέτοιες ε, συνθήκες. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από την κυβέρνηση της Κάμπιας. Σας ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Έρχομαι στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Πόλτσοκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται της αντιπολίτευσης στην χώρα αυτή. Ακόμα και μετά από τους περιορισμούς στην βοήθεια την οποία δίδουμε στις, στη χώρα αυτή και μιλάμε για 33 εκατομμύρια δολάρια παραμένουμε σαν ε, ο μεγαλύτερος δωρητής. Οπότε πώς μπορούμε να υποστηρίζουμε μια κυβέρνηση έστω και με αυτά τα ποσά. Μια τέτοια κυβέρνηση. Θυμίζω ότι το ΑΕΠ της χώρας αυτής ίσα ίσα ξεπερνάει τα 900 εκατομμύρια. Λοιπόν δεν μπορούμε να στηρίζουμε μια τέτοια κυβέρνηση, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την αντιπολίτευση και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις μόνον. Η κυρία Κιέγγε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μετά τον θάνατο του Σόλο Σαντάγκ δεν μπορούμε πλέον εμείς να ανεχθούμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι δυνάμεις καταστολής εις βάρος όλων που έχουν διαφορετική άποψη από το καθεστώς. Αρκετά στη ρητορική του μίσους, αρκετά στις εξαφανίσεις, αρκετά στις αυθαίρετες εξελέσεις, αρκετά στη λογική των πραξικοπημάτων. Ελείπει πλήρως η δημοκρατία εδώ και μάλιστα σε μια χώρα που υποτίθεται θα ψηφίσει σε λίγες μήνες οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει και στον ποινικό κώδικα, οι διώξεις εις βάρος των ΛΟΑΤ είναι καταστάσεις τις οποίες πρέπει να καταγγείλουμε. Σύμφωνα λοιπόν με τη συμφωνία του Κοτονού θα πρέπει να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν συζητήσεις με την κυβέρνηση της Γκάμπια έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε σαν παράδειγμα να δεσμεύσουμε τις πιστώσεις που προερίζονται για την Πανιούλ εκτός βέβαια από τα χρήματα που πηγαίνουν σε αυτούς που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γκάμπια είναι καθημερινό φαινόμενο. Τον Απρίλιο ξεκίνησαν οι ειρηνικέ διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Μπαντζούλ ζητώντας διαφάνεια για τις εκλογές του δεκεμβρίου του. 2016. κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτών ο ηγέτης της αντιπολίτευσης σόλο σάντεκ συνελήφθη και στην πορεία πέθανε κατά τη φυλάκισή του. στη συνέχεια υπήρξε δεύτερο κύμα διαδηλώσεων που οδήγησε σε ένα νέο γύρο καταστολής οι περιπτώσει αυτέ δεν είναι καινούργιε για την γκάμπια που αποτελεί μια από τι δεκαπέντε φτωχότερε χώρε παγκοσμίω και το ένα τέταρτο του πληθυσμού τη αντιμετωπίζει χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια. επιπλέον υπό το καθεστώ του τζαμέ από το 1994 έχουν σημειωθεί πολλές εξαφανίσεις δολοφονίες για πολιτικού λόγου και οι δυνάμεις ασφαλείας και οι παραστρατιωτικές ομάδε έχουν κατηγορηθεί για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να λάβει άμεσα μέτρα για να σταματήσει η καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην γάμπια. Ευχαριστώ. Γκάμπια είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες της Αφρικής και του κόσμου. Πάνω από το 30% του πληθυσμού ζει κάτω από το 1,25 δολάρια την ημέρα. Η ελευθερία έκφρασης δεν υπάρχει. Ε, το καθεστώς είναι ένα βίο καθεστώς, βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 20 χρόνια και πραγματικά δεν βοηθά και τους ασθενείς από AIDS, τους οποίους καταδικάζει να χρησιμοποιούν κάποια βότανα και τους καταδικάζει έτσι σε θάνατο. Ε, εφαρμόζεται φυσικά η θανατική ποινή με πάρα πολύ συχνό θα έλεγα ρυθμό. Οι διαδηλώσεις ε, καταστέλλονται και απαγορεύονται συστηματικά. Λοιπόν εμείς πρέπει εν πάση περιπτώσει να σταματήσουμε τα χρήματα που δίνουμε και να πάρουμε μέτρα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της οικογένειας του Προέδρου. Ο κύριος Ντενανό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι δεν μπορεί να αποδεχθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταπατώνται με τέτοιο τρόπο, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί ούτε και την ε, βία και τα, τους βασανισμούς στην Ζάμπια ου ή αλλού. Ο Γιαμέ έχει δημιουργήσει μια Ισλαμ... την Κάμπια σε μια ε, σε μια χώρα με Ισλαμικό δίκαιο. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει δεκτό να υπάρξει αυτή η καταπάση δημοκρατία σε αυτή τη μικρή χώρα η οποία χάνει όλο και περισσότερο τους νέους της που μεταναστεύουν για να διασωθούν. Πρέπει να παγώσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τη βοήθειά της στην Κάμπια. Αυτό δεν αφορά βέβαια τις ανθρωπιστικές ε, βοήθειες που δίνονται στην περιοχή. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον λαό, αλλά σε καμία περίπτωση τον δικτάτορα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η Επίτροπος Γιούροβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Ναι, η κατάσταση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Κάμπε πραγματικά μα ε, δημιουργεί σοβαρέ ανησυχίε, ιδίω στον τομέα τη ελευθερία τη έκφραση, των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜΑ και σε ό,τι αφορά τι αυθαίρετε συλλήψει, φυλακίσει και βασανισμού. Όλα αυτά τα αναφέρουμε με του συνομιλητέ μα, προσπαθώντα να πιέσουμε για βελτιώσει και αυτά τα θέματα είναι συχνά και στις συζητήσεις του διαλόγου του άρθρου 8 πρόσφατα στις 26 Απριλίου στην Μπαντζούλα. Οι ανησυχίε μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα έθεσαν επίσης και στις 11 Απριλίου, όταν η Εξωτερικών, ο Υπουργό Εξωτερικών της Κάμπια, είχε ε, συνομιλίες με υψηλούς αξιωματούχους στις Βρυξέλλες. Δυστυχώ, Οι καταστολές δύο ειρηνικών διαδηλώσεων 14 και 16 Απριλίου επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες μας. Οι διαδηλωτές συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν ορισμένοι και ένας πέθανε. Πολλοί εξ αυτών, ακόμη και ο ηγέτης ε, του πιο ισχυρού κόμματος αντιπολίτευσης του Ενωμένου Κόμματος, ε, δικάζονται για ε, αδικήματα μέχρι και για την και για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων ακόμη. Το Δεκέμβριο του 2016 έχουν ε, προβλέπονται εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει με δήλωσή της εκφράσει τις ανησυχίες ε, και ζητά, ζητά να διερευνηθούν τα επεισόδια σε αυτές τις διαδηλώσεις. Το ίδιο έγινε και από τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, τα Ηνωμένα Έθνη, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η οικονομική κοινότητα ε, των Δυτικών Αφρικανικών Κρατών ΕΚΟΒΑΣ ε, και η Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, ο ΙΕ, η Αφρικανική Ένωση, η ΕΚΟΒΑΣ έχουν προβεί και πραγματοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα σε μια κοινή αποστολή και εκεί ζήτησαν σεβασμό στην ελευθερία εκφρασής, στην ελευθερία του συνέχιση της πολιτικής συμμετοχής τη δίκαιη, ε, να υπάρχει δικαιοσύνη και να διερευνηθούν τα γεγονότα αυτών των διαδηλώσεων. Στην Μπαντζούλ, 26 Απριλίου, είχαμε το διάλογο του άρθρου Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε αυτό το ζήτημα ε, των, της καταστολής των ε, διαδηλώσεων. Στην Κάμπια είχε ξεκινήσει μια έρευνα και θα μας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κάμπια συνεχίζει να παρακολουθεί εκ του και στην κατάσταση, έχει επαφές με όλους τους εμπλεκομένους φορείς και ενθαρρύνει ε, στεναρά την κυβέρνηση της Κάμπια να τηρήσει το κράτος δικαίου. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε το διάλογο με τις αρχές. Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών μας και μπορεί να επηρεάσει και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη και προσιλωμένη στην υποστήριξη του λαού της Γκάμπια, στην ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και στη δημιουργία μιας κοινωνίας, ε, μάλλον μιας ε, ανάπτυξης αλληλέγγυας με βάση τις αρχές συμφωνίας του Κοτώνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε.